Προχωρούμε στις αιτιολογήσεις ψήφου. Παρακαλώ τους συναδέλφους να επιταχύνουν την έξοδό τους και να κάνουν ησυχία. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Τζουφρίντα. Κυρία Τζουφρίντα, έχετε το λόγο για αιτιολόγηση ψήφου για ένα λεπτό. Από μια έρευνα του ε, 2014 προκύπτει ότι τουλάχιστον ένας Ευρωπαίος στους 10 έχει αγοράσει αγαθές ή υπηρεσίες από τη μαύρη αγορά που προκύπτουν από αδήλωτη εργασία. Όμως ε, δεν θέλω να κάνω μαθήματα ηθικότητας ε, για η αδήλωτη εργασία είναι η Ελλάδα, στη συνέχεια είναι η Ολλανδία, η Δανία, το Λουξεμβούργο ή η Σουηδία που κανείς δεν θα τις υποψιαζόταν. Ε, μάλιστα ο κατασκευαστικός τομέας, ο τομέας των οικοδομών είναι αυτός που οργιάζει η αδήλωτη εργασία σε όλες τις χώρες. Θα πρέπει με αυτήν εδώ την πλατφόρμα να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Η πλατφόρμα λοιπόν θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα με πραγματικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Και να αναφέρω δύο μέτρα. Ε, απλοποίηση των κανόνων, χωρίς αυτό ωστόσο να θέσει ένα αμφιβόλο τις εγγύησεις και πάνω από όλα μια σημαντική μείωση του φορολογικής επιβάρησης που είναι ο βασικός ε, λόγος για την αδήλωτη εργασία. Ευχαριστώ. ευχαριστώ για ένα, το λόγο έχει για ένα λεπτό επίσης η κυρία Γκονζάλες Πένιας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι δύσκολο να ποσοτικοποιήσει κανεί τη μη δηλωμένη εργασία. Εκτιμάται όμω ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη, όπω στην Ισπανία, πλησιάζει το νούμερο στο 20% του χώριου ΑΕΠ. Και αυτό είναι τεράστιο πλήγμα για του εργαζομένου, για το κράτο, για το σύνολο τη κοινωνία. Η αύξηση τη αδήλωτη εργασία δεν έγινε τυχαία. Οφείλεται στην οικονομική κρίση και στι πολιτικέ λιτότητα, οι οποίε ε, αύξησαν την αβεβαιότητα τη απασχόληση. Και οποία βεβαιότητα πλήττει τους πιο ευπαθείς εργαζόμενους, όπως είναι οι γυναίκες, οι μετανάστες, οι νέοι και οι ψευδο ανεξάρτητοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ψηφίσαμε υπέρ γιατί είναι θετικό το βήμα για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο με συντονισμένο τρόπο. Ωστόσο, η ρίζα του κακού δεν υπάρχει. Υπάρχει και η μεταρρύθμιση στις εργασιακές σχέσεις στην Ισπανία και σε άλλες χώρες είναι μεταρρυθμίσεις που δεν θα βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος και στο ξερίζωμα του κακού, ε, το οποίο είναι η πλήρης απελευθέρωση και απορρίθμιση της αγοράς εργασίας που πλήττει τους εργαζομένους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω πως ε, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Εκατομμύρια εργαζόμενοι επηρεάζονται και πάρα πολλά κρατημέλη και η Ουγγαρία. Η πατρίδα μου, αν δούμε, σε κάθε τομέα βρίσκουμε δεκάδες χιλιάδες ε, εργαζόμενους ε, που είναι αδήλωτοι. Και οπωσδήποτε η κοινωνική ασφάλιση κινδυνεύει, πολλά έσοδα χάνονται, η ανταγωνιστικότητα επηρεάζεται επίσης. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να τονίσω πως τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και η συμπεριφορά αυτή πρέπει να τιμωρηθεί από τις κυβερνήσεις. Επιπλέον, Χρειαζόμαστε μια κοινή πλατφόρμα από τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους και το ένα με το άλλο. Ευχαριστώ. Χάναν για ένα λεπτό. Thank you, Mr. again... Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Για άλλη μια φορά ασχολούμαστε με τα συμπτώματα και όχι με την υποβόσκουσα νόσο. Γιατί πρόχνεται ο κόσμος να περάσει στην αδήλωτη μαύρη οικονομία. Γιατί η ρυθμισμένη οικονομία είναι υπερβολικά ρυθμισμένη. Οι φόροι είναι εξαιρετικά υψηλοί, οι συνθήκες εργασίες δεν είναι οι σωστές και άρα είναι συμφέρον προς τον κόσμο να δουλέψει μαύρα, να πάρει τη δουλειά του και να λειτουργήσει αλλιώς και αλλού. Η λύση δεν είναι να δώσουμε ακόμα περισσότερο φάρμακο από αυτό που δημιούργησε την νόσο και τα συμπτώματά της. Αν έχουμε ακόμα μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση, ε, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αδήλωτη εργασία. Ο όλο και περισσότεροι επιθεωρητές να αστυνομεύουν ένα σύστημα ε, θα το ε, φέρουν στα άκρα του και θα, το σύστημα θα προσπαθήσει να πάει στη μαύρη αγορά. Θα ήταν καλό να έχουμε χαμηλότερους, απλούστερους φόρους για να μην έχει κίνητρο ο κόσμος να ε, δούλεψει αδήλωτα. Έχει για λεπτό η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στηρίζω τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη βελτίωση συνεργασίας έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε την αδήλωτη εργασία. Τα δεδομένα από τις ε, έρευνες δείχνουν ότι η αδήλωτη εργασία έχει αυξηθεί κατά 20% σε ορισμένες χώρες ενώ ε, το 10% ε, δουλεύει χωρίς συμβάσεις η αδήλωτη εργασία στην Ευρώπη είναι κοινό τόπο τελικά και δεν γνωρίζουμε ποιε θα είναι οι μακροπρόθεσμε συνέπειε. Γιατί το κράτο έχει λιγότερα έσοδα και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει λιγότερα έσοδα και μειώνονται και οι συντάξεις που θα δοθούν τελικά. Επομένως, σε βάθος χρόνου θα έχουμε περισσότερους ηλικιωμένους που να διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας. Τα προβλήματα στην αγορά εργασίας προκύπτουν λόγω διαφορετικών αιτιών. Πρέπει να δράσουμε τοπικά. Και για ένα λεπτό ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Δανία έχει ένα από τα συστήματα αγοράς εργασίας που λειτουργούν καλά με μεγάλη συμμετοχή και δεν έχουμε με εκτεταμένη αδήλωτη εργασία. Δεν είχαμε τα, πρόβλημα, τα προβλήματα με που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων και υπηρεσιών. Δυστυχώς όμως ε, τα τελευταία δέκα χρόνια ε, που επιμένετε ότι ε, αυτό το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται όλο και περισσότερους κανόνες, το πρόβλημα αυξάνεται γιατί είναι δύσκολο για τις εθνικές αρχές να διώξουν όσους δεν τηρούν τους κανόνες. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερους κανόνες από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όχι. Πρέπει να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να διώκουν όσους εργάζονται μαύρα και παρέχουν μαύρη εργασία επίσης ε, σε εργαζόμενους. Πάμε σε τελείως λάθος κατεύθυνση. Για ένα λεπτό ο κύριος Μαμίκινς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια βασική αρχή του κράτους ε, δικαίου είναι η συμμετοχή του πληθυσμού στο σύστημα κατά το οποίο περιλαμβάνει τη φορολογία και τις εισφορές. Από αυτή την έννοια μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για να σταματήσουμε την αδήλωτη εργασία είναι και σημαντική και αναγκαία γιατί θα μας επιτρέψει τελικά να καταπολεμήσουμε την μαύρη οικονομία, το ξέπλυμα χρήματος και διάφορες άλλες ε, πρακτικές ε, που βλάπτουν ε, και την κοινωνία και την οικονομία. Η πλατφόρμα λοιπόν θα φέρει σε επαφή τους ειδικού των εθνικών κρατών και βεβαίως θα πρέπει να διασφαλίζονται τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων. Η πλατφόρμα δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις, είναι μια ευελικτή δομή και αυτό είναι σημαντικό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 Εγώ πιστεύω πως η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε σχέση με την ε, ε, διάδοση των πληροφοριών και των καλών πρακτικών είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να αναπτύξουμε εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να μοιραστούμε τις πληροφορίες και να επιβάλλουμε τις καλύτερες πρακτικές, να θεσπίσουμε βάσεις δεδομένων ή αλυσίδες γρήγορης αντίδρασης. Όλα αυτά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την αδήλωτη εργασία σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Και είναι πολύ σημαντικό ε, γιατί χάνουμε ε, εισόδημα, αλλά είναι το ίδιο σημαντικό και για τους ίδιους τους εργαζόμενους που πολύ συχνά είναι ακάλυπτοι, δεν ε, έχουν κανενός είδος πρόνοια και ε, γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευση. Και όσο πιο περιθωριοποιημένος είναι ο εργαζόμενος, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνουν θύματα εκμετάλλευση. Είναι σαφές ότι η, συμμετοχή και οι συστάσεις ε, για δράση είναι θελοντικά εδώ. Τέλος, ε, στήριξα την την ε, τροπολογία που λέει ότι τα μέλη δεν θα πρέπει να αποζημιώνονται για τα, ταξίδια, για τα τους έξοδα. Μπορεί δωρεάν να δίνουν το χρόνο τους και την εργασία τους, αλλά δεν είναι δίκαιο να μην πληρώνουν τα διπορικά. Já Σας ευχαριστώ. Εγώ θεωρώ πως ε, το κόστος της εργασίας είναι ε, ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο οποίο μπορούν να διακριθούν οι χώρες. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ πως θα πρέπει να διατηρήσουν τα κράτη-μέλη το δικαίωμά τους να κανονίζουν αυτά τα πράγματα εσωτερικά. Παρόλα αυτά, η μαύρη εργασία είναι πραγματικά κάτι το κακό και δημιουργεί πολλά προβλήματα, όχι μόνο στο σύστημα της ε, κοινωνικής ασφάλισης ε, και στον προϋπολογισμό, αλλά δημιουργεί πολλά κοινωνικά προβλήματα, τα ανέφεραν οι συνάδελφοι. Για τον λόγο αυτό στήριξα αυτή την έκθεση και θεωρώ πως είναι σημαντικό οι χώρες να συνεργαστούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες για να επιτήρούνται τα νόμιμα. Σας ευχαριστώ. Ε, κύριε Πόλτσακ, με συγχωρείτε, το λόγο έχει ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό. Κύριε Κέλλη, έχετε το λόγο. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί δεν μπόρεσα να μιλήσω και σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω κάτι τώρα. Πράγματι, η αδήλωτη εργασία και η μαύρη οικονομία είναι φαινόμενα πολύ έντονα σε όλη την Ευρώπη. Από 1% μέχρι και 30% ε, απαντάται το φαινόμενο αυτό, αναλόγως με τη χώρα. Το πρόβλημα προφανώς είναι τεράστιο. Ο, ο κύριος Χάναν είπε ότι ο κόσμος τίνει να δουλεύει μαύρα λόγω ε, της υπερβολικής ρύθμισης. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μικρό μέρος του προβλήματος. Ε, έμφαση πρέπει να δώσουμε στους συγκεκριμένους εργοδότες που εκμεταλλεύονται τους εργαζομένους. Χρειάζεται ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και κίνητρα ο κόσμος να πληρώσει τους φόρους του και να δηλώσει την εργασία του. Έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, μόλις προλίγου είχαμε μια συζήτηση για την αδήλωτη εργασία, δηλαδή την παραοικονομία και το Ηρωνικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά το γιατί ο κόσμος προτιμά να δουλεύει εκτός πλαισίου, εκτός κανόνων και ρυθμίσεων, ενώ ακριβώς αυτοί οι κανόνες που δημιουργούν προβλήματα εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βρετανοί συντηρητικοί και οι συνάδελφοί μου μας λένε τι καλό πράγμα που είναι η Ευρώπη και τι καλό πράγμα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είναι εφαρμόσιμη. Το Βρετανικό Εργατικό κόμμα και ειδικά στα δυτικά Midlands μιλά για ανταγωνιστικότητα και λέει θα σας διδάξουμε εμείς ένα ε, μάθημα για την ανταγωνιστικότητα. Ποιος το, λένε αυτό, ποιος το λέει αυτό οι εργατικοί που ουσιαστικά έχουν διαλύσει την οικονομία της χώρας. Όλα αυτά είναι ηρωνικά και δεν τα επινοούμε εμείς. Περνούμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση Ντέμες Μάκερ για την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοπικιλότητα. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Τζουφρίντα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Το 2015 η προσοχή στα θέματα του περιβάλλοντος ήταν πολύ μεγάλη. Το 2015 ήταν το έτος της COP21 όπου ο κόσμος αντιμετώπισε την ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας ε, του περιβάλλοντος και της φύσης. Τώρα θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένη δέσμευση μετά τη συζήτηση γιατί δυστυχώς η στρατηγική για την προστασία της βιοπικιλότητας ε, έχει αποτύχει. Ε, εκτιμώ την έκθεση της συναδέλφου που ξεκινά, από, του συναδέλφου που ξεκινά από την διαπίστωση ότι η βιοποικιλότητα είναι πόρος. Είναι πόρος και οικονομικός πλούτος αλλά και κοινωνικός πλούτος και υπογραμμίζω ιδιαίτερα την ανάγκη να προστατευτεί η βιοποικιλότητα της θάλασσας και να ενσωματωθούν οι ρήτρε για την προστασία της φύσης σε όλες τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Θα πρέπει να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα στι θάλασσέ μα και αυτό σημαίνει ανάπτυξη μέσω τη στήριξη στα πανεπιστήμια για τη μελέτη και την παρατήρηση των οικοσυστημάτων. Χωρί αυτά ο κόσμο θα είναι φτωχότερο και η υγεία μα ε, χειρότερη. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Στήλερ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσο φιλελεύθερη θέλω να προστατεύσω την οδηγία αυτή. Δεν θα πρέπει να είναι δικαιολογία για να αποδυναμώσουμε την νομοθεσία. Πρέπει η μείωση της γραφειοκρατίας να μην είναι δικαιολογία για να ε, πλήττεται η βιοποικιλότητα και το περιβάλλον πρέπει να γίνεται δημόσια διαβούλευση για τα ωφέλη της οδηγίας. 100.000 πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο μίλησαν υπέρ της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Στη Σκοτία έχουμε το Nature Science και όλα αυτά τα μέρη προστατεύουν την χλωρίδα και πανίδα. Δηλαδή το ότι οι περιοχές στη Σκοτία έχουν μπει στο δίκτυο Natura. Ως προς τα πτηνά, Έχουμε 153 ε, ζώνες ειδικής προστασίας. Είναι τεράστιος ο αντίκτυπος για τη διάσωση της βιοπικιλότητας στη Σκοτία. Θέλουμε να εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Μαμίκινς. Σας ευχαριστώ. Ένας υπεύθυνος ε, ιδιοκτήτης ε, φροντίζει ώστε η περιουσία του να είναι σε καλή κατάσταση, καθαρή και από καιρού εις καιρό κάνει απεντόμωση. Ε, οι ιδιοκτήτες τέτοιου τύπου μπορεί να θεωρηθεί ε, ότι είναι ιδιαίτερα ανθρωποκεντρική θα έπρεπε και εμεί να φροντίζουμε με τον ίδιο τρόπο τη φύση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως η γη μας είναι το μόνο μας σπίτι. Δυστυχώς ε, οι σημερινέ τάσει σημαίνουν ότι δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους ε, στην Ένωση για βιοποικιλότητα μέχρι το 2020. Θα έπρεπε να υπάρχει ε, μια ενδιάμεση αξιολόγηση, αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, συνεργασία ανάμεσα στις διεθνείς και τοπικές δομές, καθώς και κοινή γεωργική πολιτική και κοινή αλευτική πολιτική. Ευχαριστώ. Um, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο παρότρινε τα κράτη-μέλη να μην εγκρίνουν οποιαδήποτε ε, νέα διαδικασία υδρορογμάτωσης στην Ένωση και αυτή η έκκληση έγινε επί τη βάση της αρχής της προφύλαξης αλλά και λόγω των κενών της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που διαπιστώθηκαν. Είπαμε ότι χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τους κινδύνους και το αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα και στη βιοπικιλότητα καθώς και στο περιβάλλον που ε, περιέχεται στην υδρορογμάτωση και σε αυτή τη διαδικασία. Ε, υποστηρίζουμε αυτή την ε, ιδέα, αυτή την άποψη και με ξέπρεξε κάπως το ότι χρειάστηκε να αντιπαρατεθώ με τους συναδέλφους στο Sligo County, στην κομιτεία του Sligo, γιατί δεν θέλησαν να ακολουθήσουν αυτήν την ε, γραμμή, είναι ένα σχέδιο και ίσως να μπορεί να αλλάξει. Ε, ίσως όμως ε, η σημερινή ψηφοφορία εδώ να επηρεάσει και τα αποτελέσματα εκεί στην Ιρλανδία. Για ένα λεπτό ο κύριος Μπέντσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι υπέρ της έκθεσης αυτής που έτυχε ευρεία πλειοψηφία. Στο άρθρο 68 στηρίζουμε την εξή αρχή, ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι ε, λεπτομερείς. Ξέρετε, η φύση δεν είναι ένα στατικό φαινόμενο και δεν θα πρέπει να είναι και η δράση μας στατική. Ξέρετε, παλιά η λύκη ήταν επαπειλούμενο είδο. και σήμερα όμω δεν είναι πια. Πρέπει να ρυθμίσετε αυτό το θέμα εθνικά. Το λόγο έχει για ένα λεπτό επίσης ο κύριος Πόλτσακ. Σας ευχαριστώ και εγώ ήμουν υπέρ αυτής της ε, έκθεσης ε, γιατί η ποικιλομορφία είναι βασικό σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η βιοπικιλότητα είναι επίσης σημαντική στην Ήπειρό μας. Είναι σαφές πως η στρατηγική μέχρι στιγμής δεν ήταν πολύ επιτυχημένη και πρέπει να αντιληφθούμε πως η βιοπικιλότητα δεν ε, είναι μόνο θέμα του περιβαλλοντος. Η προστασία της ε, φύσης είναι βασική αξία, αλλά είναι και ένα κοινωνικό στοιχείο εγώ δεν είμαι υπέρ των υπερβολικών κανόνων. Μιλάμε συχνά για μια τροφία που δημιουργεί το δίκαιο, όμως το περιβάλλον είναι ένας τομέας που πραγματικά αξίζει να έχει σωστούς κανόνες ε, για τις επόμενες ε, γενιές. Μπορούμε βεβαίως ε, πράγματι να καταπλούμε τα ευλαβία, να αναφήσουμε και κλονίες επόμενες γενιές. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή που επέμεινε στο γεγονός ότι η βιοπικιλότητα είναι κάτι το ε, πολύ σημαντικό και ότι είναι επίγον να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση κυρίως ε, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους για το 2020 αλλά και τα αποτελέσματα της διάσκεψης των μερών ε, για το κλίμα 21 που έλαβε χώρα στο Παρίσι υπονομεύεται, υποβαθμίζεται η βιοπικιλότητα συνεχώς και οφείλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Όχι μόνο όλοι μας, αλλά και κάποιοι οφείλουν να κάνουν πολύ περισσότερα από ό,τι έκαναν πριν και πολύ περισσότερα από τους υπόλοιπους. Θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν ε, τα ωφέλη αυτού του εγχειρήματο. Ξέρετε, στην περιοχή όπου ζω, ε, Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ακούσαμε και τον Εστονό Πρόεδρο. Ήταν πολύ συγκεκριμένος και τα λόγια του με βρισκούν απολύτως σύμφωνο. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε την αιτιολόγηση ψήφου. Η συνεδρίαση διακόπτεται έως τις 3 το απόγευμα σήμερα. Σας ευχαριστώ. Είμαστε μια